Και πέρα από αυτό εμείς ως Επιτροπή ε, είμαστε υπόλογοι για κάθε μέτρο ενώπιον του Κοινοβουλίου. Στη φάση αυτή, μετά την ανταλλαγή με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και μετά την ε, διαβούλευση, της για την έκθεση, θα πρέπει να συζητήσουμε εις βάθος τα εξής θέματα. Τη σχέση μεταξύ λήψεων και οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, άρθρο 7. Η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει γκρίζα ζώνη μεταξύ διαφόρων οργάνων και δυνατοτήτων ανάληψης ε, δράσης. Εδώ έχουμε τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες, οι οποίες θα επαγρυπνήσουν ούτε ώστε τα πάντα να διατυπωθούν απολύτως ξεκάθαρα ποιο όργανο, σε ποια περίπτωση, ε, ποιο εργαλείο, σε ποια περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ε, και θα πρέπει οι ελλείψεις στις χώρες μέλη να είναι να διατυπώνονται με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο. Ο κατάλογος σας των ελλείψεων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος, αλλά θα πρέπει να είναι ανοιχτός για να μπορεί ο μηχανισμός να εφαρμοστεί και σε απρόβλεπτες ε, περιστάσεις και καταστάσεις. Υπάρχει μια ενδεικτική προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να λαμβάνει γνώση η Επιτροπή Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό περιθώριο αλλά είναι σημαντικό η Επιτροπή να κάνει μια, έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει το χρονικό αυτό περιθώριο που έχει στη διάθεση της Επιτροπή να είναι υπερβολικά περιορισμένο. Επιθυμούμε να μελετήσουμε τις ε, ε, επιθυμούμε να διευκρινιστούν συγγνώμη, οι πηγέ πληροφόρηση ε, στι οποίε θα βασίσει την εξολόγησή τη η Επιτροπή. Ο κατάλογο τη νομολογία στι οποίε μπορεί να βασιστεί η Επιτροπή, καθώ και οι πηγέ ε, πληροφοριών που μπορούν βεβαίως να κοινοποιηθούν και στο Κοινοβούλιο. Επίσης το ερώτημα δεν κάνεις λίγο κουράστηκα. Ο μηχανισμός του κράτους δικαίου που συζητάτε σήμερα και που νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια εδώ, αποτελεί σημαντικό οικονομικό λίθο για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα καλύψει το διάστημα 2021 έως 2027. Θα πρέπει να υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή, ώστε ο προϋπολογισμός να μπορέσει να συμβάλλει στην προστασία των ε, φόρων που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Έτσι συμπληρώνουμε ένα κενό στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας καλώ λοιπόν να συμπληρώσετε το κενό αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να φροντίσετε να έχουμε εντός του έτους μια απόφαση που θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τον προϋπολογισμό της επόμενης δεκαετίας. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μιχαήλοβα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στη γνωμοδότησή της για την έκθεση αυτή ε, επισημαίνει ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, είναι υψής της σημασίας για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε απόφαση για την εφαρμογή μέτρων σε περίπτωση γενικευμένων ελήψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου θα πρέπει να υπάρχουν σαφή εχέγγυα σε μια μελέτη αντικτύπου ώστε να φροντίσουμε οι ε, τελικοί δικαιούχοι των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να μην ε, θίγονται. Το εύρος και το επίπεδο των κυρώσεων θα πρέπει να είναι αναλογικό και θα πρέπει να βασίζεται στην ίση μεταχείριση των κρατών μελών και να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στο κράτος μέλος. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου, μπορεί να εφαρμόζεται και ο κανονισμός ε, ε, γενικών διατάξεων για να προστατευτούν οι τελικοί δικαιούχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη, να φροντίζει όμως επίσης ε, οι θεσμοί των κρατών μελών να εκταμιεύουν τα σχετικά ποσά. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Σόλς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, στο όνομα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ε, τονίζω ότι είναι σημαντικό ε, να προστατεύουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη. Ναι, υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτή την πρόταση και την εκτέλεση του προπολογισμού ε, σύμφωνα με τι αρχέ τη καλή δημοσιονομική διαχείριση είναι απαραίτητο να ε, φροντίζουμε για την εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου. Γι' αυτό η Επιτροπή ΑΦΚΟ προτείνει ε, ε, προς όφελος τη δημοσιονομική αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη να διασφαλίσουμε την συνεργασία των κρατών μελών προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει οι ε, τελικοί δικαιούχοι των ε, προγραμμάτων ή των ταμείων να μην θίγονται από τις κυρώσεις αυτές. Και γι' αυτό προτείνουμε αξιολόγηση των εθνικών προϋπολογισμών και τέλος πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρα από το δικαίωμα της ενημέρωσης, ε, θα πρέπει ε, να έχει ισχυρό ρόλο όσον αφορά την αξιολόγηση της διαδικασίας. Ε, θα πρέπει να είναι διαφανής η σχετική διαδικασία. Πολιτικών ομάδων, για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει η κυρία Γκρέσλε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, συνάδελφοι. Οχτώ άρθρα ε, έχει η πρόταση αυτή, αλλά ε, τρέφω πολλές ελπίδες όσον αφορά τα άρθρα αυτά, διότι είναι ο πρώτος ε, κανονισμός που ασχολείται με τις γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Επικροτώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την έκθεσή τους. Είναι σημαντική αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη με διεφθαρμένες δομές. Βλέπουμε εκπροσώπους κυβερνήσεων που εκμεταλλεύονται την επιρροή τους ως επικεφαλής των κυβερνήσεων ώστε να φροντίζουν οι ίδιοι οι φίλοι τους ε, να λαμβάνουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να υπάρχουν λύσεις. Ε, μια διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 δεν θα λύσει το πρόβλημα αυτό, διότι ε, στο άρθρο αυτό προβλέπεται μια γενική δικαστική διαδικασία, ενώ τώρα μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που γεμίζουν τις τσέπες τους και κλείνουν το στόμα στους δημοσιογράφους. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να εξετάζουμε τι γίνεται σε περίπτωση απάτης και νομοποίησης ε, παράνομων ε, εσόδων, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πρέπει να εξοραγήσουμε την κατάσταση. Ο κανονισμός αυτός δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει έναν τρόπο να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις. Θα είναι θετικό αύριο να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Και δημοκρατών, το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Γιάλα Σέντερ. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Γκαρσία Γουαρδία Σαμπάλα αλλά και τον κύριο Σερβάμα για τη δουλειά που έχουν κάνει σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Είναι, πραγματικό, είναι αλήθεια ότι θα, θα προτιμούσαμε άμεσες ε, κυρώσει και πολιτικέ από το Συμβούλιο και να μην έρχεται στην Κομισιόν και στο Συνοβούλιο να ολοκληρώσουν μια εργασία που τελικά επηρεάζεται πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ε, Πάντως οι δύο εισηγητές ε, κατάφεραν να φτιάξουν ένα καλό κείμενο όπου ε, προστατεύονται πραγματικά τα κονδύλια γιατί αν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη αν δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν μπορούν να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ταμείων που επηρεάζουν τη ζωή ε, των δικαιούχων, των πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις συνήθειες των κυβερνήσεων μέσω οικονομικών κυρώσεων. Πρέπει λοιπόν οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται από τους ε, πολιτικούς υπεύθυνου ε, ε, ώστε να μην καταλήγουμε σε κίνδυνο και σε ε, αντιπαράθεση. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε αυτό εδώ να το ολοκληρώσουμε πολύ πιο γρήγορα. Ήταν καλό το κείμενο, δύσκολο και περίπλοκο, αλλά αν καταφέρουμε να το εφαρμόσουμε και να το εξηγήσουμε καλά, θα καταφέρουμε αυτό που είναι ο στόχος μας, ότι δηλαδή για να καταφέρουμε να έχουμε αυτή την Ευρώπη που προστατεύει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε προστατεύοντάς την από αυτούς που θέλουν να την ζημιώσουν. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω τα καταφέραμε καλά. Όχι, κινέζικα. <laughs> Να το. Στόπα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους, με με τη συνάδελφα κυρία Γιάλα Σάντερ, θα πρέπει να προστατεύσουν την Ευρώπη από αυτούς που θέλουν να την καταστρέψουν. Το ερώτημα είναι ποιος επιθυμεί να καταστρέψει την Ευρώπη. Εκείνοι που πυροδοτούν ε, το κύμα ευρωσκεπτικισμού στις χώρες μέλη ή εκείνοι οι οποίοι παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των χωρών μελών ή εκείνοι που ανθίστανται είτε στις κάλπες είτε στους δρόμους, γιατί αυτό το είδαμε σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Αυστρία, τη Τσεχία, την Πολωνία, την Ουγγαρία. Ο κύριος Σάρβαμα έχει... είχε δίκιο όταν μίλησε, αναφέρθηκε στο κουτί της Πανδώρας, αλλά δεν θα έπρεπε να ανοίξουμε αυτό το κουτί με τέτοιου διατάξεις οι οποίες μπορούν να παρερμηνευθούν. Η χώρα του Επιτρόπου κυρίου Έτιγκερ έχει βεβαίως ε, το δικαίωμα να επιλέγει τον πρόεδρο του συνταγματικού δικαστηρίου στην Καλσρούη. Δεν θέλουμε να ανακατευθούμε στα εσωτερικά της Γερμανίας, αλλά θα πρέπει να ισχύει και το αντίστροφο. Ε, τέτοιες ε, χώρες που, ε, σε οποίες γίνεται επίθεση όπως η Ουγγαρία, ε, έχουν αποφασίσει δημοκρατικά για τον τρόπο διακυβέρνησής τους. και Δημοκρατών, το λόγο έχει η κυρία Μάκη για λεπτό. Η αρχή του κράτους δικαίου είναι η βάση για όλες τις δημοκρατικές χώρες. Εάν δεν κατοχυρώνεται η αρχή του κράτους δικαίου, τότε παρεμποδίζεται και η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών καθώς και η διαβίωση των πολιτών. Όταν μια χώρα προσπαθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να εκπληρώσει συγκεκριμένα κριτήρια. Εδώ πρόκειται για ανάληψη μια κοινή ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόταση αυτή δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματα. Εδώ έχουμε πολύ ψηλέ προσδοκίες, αλλά η πρόταση αυτή αφορά την προστασία όσον αφορά τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, ασφάλεια, την εξασφάλιση ότι χρησιμοποιούνται ε, σωστά τα κονδύλια αυτά. Αλλιώς η διαδικασία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Άρα λοιπόν το εργαλείο αυτό δεν ε, επιλύει το πρόβλημα με γενικότερους όρους όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου στις χώρες μέλη. Και δεν είμαι σίγουρος ότι η εφαρμογή του μηχανισμού αυτού ε, στην πράξη θα είναι επιτυχής. Εμείς ε, προτείναμε μεν κάποιες βελτιώσεις, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε την προστασία των τελικών δικαιούχων. Η δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζει αυτή την πρόταση, αλλά από νομική άποψη ο κανονισμός αυτός είναι μάλλον πολύπλοκος και γραφειοκρατικός. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. έχει για δύο λεπτά η κυρία Νιρίντα. Πρέπει να σας πω ότι αφού διάβασα το έγγραφο Έχω κάποιες ανησυχίες ε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς και ακόμα και αν μιλάμε για το κράτος δικαίου, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι το μετατρέπουμε σε πολιτικό μέσο. Είναι δύσκολο λοιπόν να εφαρμοστούν οι κανόνες προς τη μια κατεύθυνση και μετά προς την άλλη. Ε, πιστεύω πως θα υπάρχουν πλεονεκτήματα για τις πλούσιες χώρες, για παράδειγμα, ε, και έχω την εντύπωση πως ε, δημιουργούμε μια κατάσταση όπου οι χώρες δεν θα είναι υπεύθυνε για τα χρήματα που ε, εισέρχονται στις χώρες τους, αλλά εμείς πρέπει να προστατέψουμε τον προπολογισμό μας. Πιστεύω πως η Κομισιόν δεν θα πρέπει να έχει τέτοιο επίπεδο αρμοδιότητας και εξουσίας να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου σε ορισμένες χώρες. Η Κομισιόν κάνει πίσω όταν βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ισπανία και την κατάσταση κατάσταση στην Καταλωνία όταν θέλουν να ψηφίσουν η Κομισιόν κάνει πίσω και δεν λέει τίποτα για αυτούς που επιθυμούν ε, να γίνει ψηφοφορία. Αλλά τώρα έχουμε μια απόφαση και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ισότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Μιλάμε για εμπορικά ζητήματα. Ε, Βλέπουμε ότι υπάρχουν πλανεκτήματα για όσους ε, τα με την Κομισιόν. Χρειάζεται ε, σαφήνεια, χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Νομίζω πως αυτές οι χώρες που ήδη υποφέρουν δεν θα, δεχτού, δεν θα λάβουν ε, την απαραίτητη βοήθεια. Θα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει πολιτικά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το μεγάλο θέμα στη συζήτηση αυτή είναι υπό ποιες προϋποθέσεις θα χρησιμοποιείται το μέσο αυτό. Διότι αν μιλάμε για κατάχρηση ε, ταμείων ε, και κακή χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων, αυτό είναι ένα θέμα και ε, κανείς δεν θα είναι πιο αντίθετος από μένα στην λάθος χρήση των πόρων. Αλλά ε, αν ε, μιλάμε για περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι κάποιος έχει ενεργήσει με τρόπο που δεν της αρέσει και ουσιαστικά λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις εις βάρος κάποιου κράτους μέλους, αυτό είναι άλλο θέμα και νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Σανάκη. Εμένα με απασχολεί η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όπου ε, το Συμβούλιο ε, έχει μόνο τη δυνατότητα να αντιδράσει με αρνητική ειδική πλειοψηφία. Μου φαίνεται ότι είναι λάθος η κατεύθυνση. Αντίστροφα θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να υποβάλει κανείς αποδεικτικά στοιχεία ότι κάτι πάει στραβά και όχι απλά να πρέπει να ανατραπεί μια σχετική απόφαση. Και φοβάμαι ότι έτσι οδηγούμεθα σε μια κατάσταση όπου έχουμε την μη εκλεγμένη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπαγορεύει στις κυβερνήσεις ε, τι να κάνουν. Και φοβάμαι ότι δεν ε, θα ισχύει η ίδια διαδικασία Είτε μιλάμε για την Ισπανία είτε μιλάμε για την Πολωνία. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα είναι πολιτικοποιημένη η διαδικασία και κύριε Πρόεδρε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δείξει ότι είναι προσιλωμένη στο κράτος δικαίου, θα πρέπει να μιμηθεί τις βέλτιστες πρακτικές όσων ακολουθούν το κράτος δικαίου και μου φαίνεται ότι λείπει το στοιχείο αυτό από την πρόταση αυτή για την ομάδα των Εθνών και της Ελευθερίας. Το λόγο έχει ο κύριος Ζόουτεκ για 1,5 λεπτό. <clears throat> Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι το τελικό βήμα για να αναλάβει την εξουσία των κρατών μελών. Από σήμερα μπορούν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να περικόψουν τις ε, επιδοτήσεις προς τα κράτη-μέλη. Ε, και δεν αρκεί τώρα πια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ισότητα στα κράτη-μέλη, η αναγνώριση των ομοφιλόφιλων ή το θέμα των προσφύγων. η πολωνική οικονομία ε, τα επόμενα χρόνια θα καταστραφεί από ε, τέτοια μέτρα. Και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την τελευταία λέξη. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει το κίνημα Paul Exit για να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο Ρόμπερτ Σούμαν προέβλεπε ελευθερία μετακινήσεων ε, σε μια Ενωμένη Ευρώπη, αλλά μέχρι εκεί. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε τη χώρα μας απικία και να την ε, ξεζουμίζεται, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Σας καλώ να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη όπως είχε προβλεφθεί αρχικά ή να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγραμμένος. Το άρθρο 3 της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Η αρχή της κυριαρχίας εδράζεται στο έθνος. Ε, κανένα σώμα το κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκήσει ε, άλλο είδους εξωσυσία δίδοντας ε, στους επιτρόπους ε, δυνατότητα επιβολής ε, κυρώσεων έναντι χωρών μελών που δεν σέβονται τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζεται η ελευθερία, απόφαση εκ μέρους των πολιτικών για τη χάραξη της πολιτική τους. Για παράδειγμα, η άρνηση του κυρίου Ορμπάν να ανοίξει τα σύνορά του σε όλους τους αθλίους του κόσμου. Ε, σε αυτό θέλετε να επιβάλλετε κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ανακυκλώνει ε, ένα αυθαρχικό μοντέλο υπό το πρόσχημα της δημοκρατικότητας ε, γιατί ζήτω η λαϊκή κυριαρχία, ζήτω η δημοκρατία. Για 1,5 λεπτό κύριος domnule ε, președinte, ε, stimați colegi. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ ότι έχουμε ανάγκη αυτού του κανονισμού. Ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και όλοι οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Εάν μια χώρα μέλος δεν ε, σέβεται μία από τις ε, αρχές του κράτους δικαίου, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση και προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Ε, προτείνει κάποιες ε, διευκρινήσεις στην πρόταση της Επιτροπής. Υπάρχουν όμως και άλλες ελλείψεις. Δεν υπάρχει επαρκής ε, διατύπωση όσον αφορά τον τρόπο που οι ελλείψεις ε, όσον αφορά το κράτος δικαίου επηρεάζουν τον προπολογισμό. Και δεν υπάρχουν αρκετές εγγυήσεις ότι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων θα λάβουν τα χρήματά τους σε περίπτωση που υπάρξει αναστολή ε, της εκταμίευσης προς τις χώρες αυτά, αυτές. Ε, υπάρχει διαδικασία του άρθρου 7. Εγώ ελπίζω οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα καταλήξουν να καταργήσουν αυτές τις ασάφειες ούτως ώστε να έχουμε επιτέλους ένα κανονισμό ο οποίος να μπορεί να ωφελεί τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η δημοκρατία είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο και εύθραυστο κόσμημα και πολύ σοβαρό για να την αφήσουμε στο έλεος των κυβερνήσεων. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς κράτος δικαίου, ε, όπως το αναφέρει το προήμιο της Χάρτας των Μολεμών Δικαιωμάτων. Η Ευρώπη δράζεται στην αρχή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αναφέρει. Άρα λοιπόν έχει το καθήκον να την εγγυάται. Ωστόσο τα τελευταία αυτά χρόνια η οι ε, παρεκκλήσεις, που είναι απαράδεκτες ε, έχουν αναδυθεί όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, την εξαρτησία της δικαιοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και δυστυχώς ε, πολλαπλασιάζονται σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Και θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Ε, κα, ε, καμία χώρα δεν βρίσκεται στο απειρόβλητο. Άρα είναι κατεπήγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις και να στραφεί κατά των ενόχων κυβερνήσεων. Εμένα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρωτοβουλία, ιδιαίτερα τους συναδέλφους και ιδιαίτερα όμως τους συναδέλφους ε, κυρία Γκαρθιαμπάλ και Σαρβανά όσον αφορά τη δημιουργία αυτών των ε, μηχανισμών καλύπτοντας ένα έλλειμμα του νομικού μας συστήματος, όπως είπε ο Επίτροπος κ. Σέτιγκερ. Ωστόσο, ε, θα πρέπει να υπάρχει μια νομική ε, βάση για το μηχανισμό αυτό και θα πρέπει να προσθεθεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ε, κάτι που θα πρέπει να μας κρούσει τον κόδωνα κινδύνο σε αυτή την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και για δύο λόγους. Το πρώτο όσον αφορά την εφαρμογή για να ελέγξουμε ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται στις κυβερνήσεις και όχι στους πολίτες δικαιούχους. Γιατί θα ήταν παράλογο να είναι οι φοιτητέ, τα ερευνητικά εργαστήρια, τα πανεπιστήμια, οι γεωργοί ή οι περιφέρειες που να είναι θύματα σφαλμάτων που έχουν διαπράξει κυβερνήσεις γιατί πραγματικά αυτή θα ήταν μια διτή ποινή. Επίσης θα πρέπει να επαγρεπνήσουμε το ώστε να εμποδίσουμε ένα τέτοιο είδους εργαλείο υπεράσπιση των αρχών του κράτους δικαίου να μην εκφυλιστεί σε εργαλείο ε, διαχείρισης του προπολογισμού ή διαχείρισης της ε, ένδυας του προπολογισμού ε, βλέποντας ακριβώς τη φτώχεια του προπολογισμού μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι παρότι οι εισηγητές θα έπρεπε να καθορίσουν τα κριτήρια για τις ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, παρόλα αυτά έχουν αφήσει μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας. Αυτό αντιστοιχεί και στην ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι και οι, οι υπάρχουσες διατάξεις μας επιτρέπουν ε, να μπλοκαριστούν οι πόροι όταν ε, δεν εφαρμόζεται δημοσιονομική πειθαρχία. Έχουμε το παράδειγμα της ε, Γαλλίας και του υπερβολικού δημοσίου χρέους. Η Γαλλία δεν τιμωρήθηκε. Τα νέα λοιπόν αυτά μέτρα τα οποία μπορούν να ε, επιβάλλονται αυθαίρετα είναι ε, ανεύθυνα μέτρα και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, για να προστατευτεί ο προπολογισμό τη Ένωση και τα οικονομικά τη συμφέροντα για το επόμενο PDP, χρειάζεται ένα κανονισμό που να μην είναι τιμωρητικό, αλλά που θα εξασφαλίζει την ορθή διαχείριση άρθρο 2 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη, στα, στοιχεία, στα κριτήρια της Κοπεχάγης ε, ε, υπάρχουν όλα αυτά. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, μπορεί αυτό να επηρεάσει την ορθή οικονομική διαχείριση και να επηρεάσει ή να ζημιώσει τα συμφέροντα της Ένωσης. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένα σύνολο, να, να, να συγκληθεί ένα σύνολο εμπειρογνωμόνων που θα εκτιμά την ε, κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και όταν θα λαμβάνει η Κομισιόν τις αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ε, γνωμοδότηση της συγκεκριμένης ε, ομάδας. Επίσης η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οτιδήποτε οφείλουν οι κρατικοί οργανισμοί, τα κράτη-μέλη θα καταβάλλεται στους δικαιούχους. Το Κοινοβούλιο τίθεται δε επίσης όρισε με το Συμβούλιο στη διαδικασία έγκρισης ή ε, κατάργησης των ε, λόγων μέτρων. Η Κομισιόν προτείνει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο τη μεταφορά των αποθεμάτων μόνο ε, και αυτό θα γίνει μόνο εάν το εγκρίνουν και τα δύο όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή την πρόταση είναι να καθοριστεί η χορήγηση των κονδυλίων προς τα κάτι μέλη με προϋπόθεση του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου όμως ποιος θα το ορίσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση η Κομισιόν είναι αυτή που θα ελέγξει τα κράτη-μέλη, αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αρνήθηκε τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στην Ιρλανδία, την Ολλανδία και τη Γαλλία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αυτή η Ευρωπαϊκή Κομισιόν που δεν δέχεται το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου όπου ο Κόσμο ελεύθερα επέλεξε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθεί την ανακεφαλοποίηση του οικονομικού συστήματο με τα δημόσια χρήματα και μετά υποβάλλει το λογαριασμό στους λαούς με την πολιτική ε, λιτότητα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αφήνει να πνίγονται χιλιάδες στη Μεσόγειο και που τους κάνει, ε, τους μεταχειρίζεται σαν εγκληματίες. Ε, ο κατάλογος αυτός δεν ε, έχει τέλος. Λείπει η νομιμοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγχει το κράτος δικαίου. Οι λαοί τη Ευρώπη θα πρέπει ελεύθερα να επιλέγουν το μέλλον τους, να επιλέγουν πόσο και αν θα αναπτυχθούν και πάλι αυτό το μοντέλο θα πρέπει να το διαγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, απορρίπτουμε λοιπόν κάθετα αυτό το μέσο. Voorzitter, Vandaag Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε σήμερα για την προστασία του προπολογισμού τη Ένωση στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη. Όπω καταλαβαίνετε από τον τίτλο, Μα ενδιαφέρουν τα χρήματα, αυτά που δαπανώνται για παράδειγμα στην Ουγγαρία ή την Πολωνία, ενώ δεν πληρούν τα κριτήρια, δεν εφαρμόζουν τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν το νέο μέσο στόχο έχει να εμποδίσει τη χρηματοδότηση για τις χώρες αυτές. Ε, θα πρέπει να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη όσον αφορά τη φορολογία, γι' αυτό θα έχουμε ανεξάρτητη αξιολόγηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή σε κάτι που θα υπονομεύσει περαιτέρω την κυριαρχία των κρατών μελών. Το εργαλείο αυτό στόχο έχει την ε, Πολωνία και την, Ουγγαρία, τις περήφανες αυτές χώρες ε, που ε, πρόσφατα βγήκαν από δεκαετίες δικτατορίας. Εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση. Αξιότιμη εκπρόσωπε της Επιτροπής, από τη συνάδελφη, με εντυπωσιάζει η κατεύθυνση προς την οποία κινείται η συζήτηση. Ένα είναι ξεκάθαρο. Τα, ε, οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δώρο, αλλά επενδύσεις. Και αν ε, σε κάποιες χώρες η καταπολέμηση της απάτης για τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν λειτουργεί, θα πρέπει να γίνει κάτι. Για παράδειγμα, 80% το 2017 δίδονται από τις ε, χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουν, εάν υπάρχει απάτη, να λαμβάνεται δράση. Χώρες όπως η Πολωνία το 2016 πήραν 10,6 εκατομμύρια, η Σλοβακία 2 δις, η Ουγγαρία 5 δις ε, κλπ. Και οι χώρες αυτές πραγματικά παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα με την πρόταση αυτή ε, η Επιτροπή επιτέλους θέλει να παγώσει ή να αναστείλει την εκταμείευση πόρων ε, μέχρι να αποκατασταθεί τάξη. Η, ε, τα κονδύλια είναι συνδεδεμένα με κάποιους όρους. Δεν είναι δώρο, είναι επενδύσεις και όταν ε, δεν αλλάζει η συμπεριφορά των παραληπτών θα πρέπει να υπάρξουν επιπτώσεις γιατί όταν ξοδεύονται χρήματα των φορολογουμένων ε, και πάνε σε κάποιες χώρες θα πρέπει οι χώρες αυτές να τηρούν τους κανόνες. κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τους Ευρωπαίους πολίτες να σέβονται τις αρχές και τις αξίες της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εάν οι ίδιοι που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους είναι τα κράτη-μέλη και αν και χάρη σε μια κοινή κουλτούρα του κράτους δικαίου, τα πλευρά των ε, θεσμών μπορούμε να ε, πιστοποιήσουμε και να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εγγυηθούμε την εκτέλεση των πολιτικών. Γι' αυτό αυτές οι γενικευμένες ελλείψεις που αφορούν το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη και που έχουν αντίκτυπο στην ε, ορθή ε, ε, οικονομική διαχείριση της Ένωσης θα πρέπει να βρουν αντίθεση όχι μόνο για να εγγυηθούμε τα συμφέροντα της Ένωσης αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινή γνώμης στην Ένωση και στους θεσμούς. Δεν καταλαβαίνω τι κρύβεται πίσω από τις τροπολογίες κατάργησης της πρότασης της Κομισιόν. Αντίθετα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να εγγυηθούμε το σεβασμό ε, και την προώθηση των αξιών και των αρχών και των δικαιωμάτων καθώς και την ομιμότητα του ευρωπαϊκού project για μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες. Ευχαριστώ. Λόγο έχει η κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ένωση χαρακτηρίζεται από κοινέ αρχές και αξίες και ενώ Κανείς δεν θέλει να του υπαγορεύουν πώς ε, να κάνει τα πράγματα προς ε, δικό του όφελος. Ε, οι θεμελιώδεις αξίες θα πρέπει να εφαρμόζονται. Είναι λοιπόν σωστό τα κράτη-μέλη που παραβιάζουν τις αρχές αυτές να μην έχουν το, πρόσβαση στους κοινούς οικονομικούς μας πόρους. Ωστόσο, άλλα λέει η θεωρία, άλλα λέει η πράξη. Έχουμε δει πολύ ε, περίεργες ε, ε, ε αρχές ε, όσον αφορά τις κυρώσεις κρατών μελών που δεν ακολουθούν τις κοινέ αρχές. Εγώ θέλω να καταλάβω τι σκοπούς εξυπηρετούν οι μηχανισμοί αυτοί και γι' αυτό θα καταψηφίσω την έκθεση. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πλειοψηφία των ευρωσκεπτικιστών ε, βουλευτών θα έρθει εδώ ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ενισχύσει τις αρμοδιότητές της καταστολής. Τελευταία αυτή η απόπειρα είναι να ε, ε, καταργηθεί η χορήγηση χρηματοκοδηλίου στα κάτι μέλη που υποτίθεται δεν έχουν το κάτω δικαίωμα. Δηλαδή μπορεί να, κόψει, να, να κλείσει την κάνουλα σε οποιαδήποτε χώρα δεν ε, υπακούει στη δικά τη καπρίτσια. Είτε πρόκειται για μετανάστε, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Αυτή ο μόνιμο εκβιασμό για τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι απαράδεκτος, γιατί ακριβώ αυτά τα κονδύλια προέρχονται από τις συμβολές των κρατών μελών και γιατί αυτές οι κυβερνήσεις, Ιταλική, Πολωνική ή η η που τόσο δυσαρεστούν την, Ένωση, την Κομισιόν έχουν εκλογεί από τους λαούς αυτοί ε, και γι' αυτό και απορρίπτουμε κάθε είδους αιρεσιμότητας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για 1,5 λεπτό. Ε, ε, Csodálkozva Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται να υπάρχει θεσμικός φετιχισμός κάτι που με εκπλήσει. Φαίνεται ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων ε, να είναι η διασφάλιση του κράτους δικαίου. Συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εστιάζουν στη διασφάλιση της ελευθερίας των Ευρωπαίων πολιτών. Και να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε ε, να διασφαλίζεται η ευημερία της Ευρώπης, η διασφάλιση της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας. Αυτά μας βοηθάει το κράτος δικαίου να πετύχουμε. Η νομοθεσία, τα θεσμικά όργανα, οι κανόνες εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Φυσικά, υπάρχουν διάφορα φαινόμενα τα οποία απειλούν το κράτος δικαίου. Ό,τι και να γίνεται όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται να υιοθετεί απόφαση με την οποία να υιοθετεί μέτρα που να παραβιάζουν το κράτος δικαίου στο όνομα της προστασίας του κράτους δικαίου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ασθενής, αποδυναμώθηκε περαιτέρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν καθορίζεται με ακρίβεια η διαδικασία για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Η πρόταση αυτή αντίκειται στο κράτος δικαίου και γι' αυτό δεν τη στηρίζουμε, ούτε και εσείς θα πρέπει να τη στηρίξετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί μιλάμε και πάλι για το κράτος δικαίου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συγκινεί ε, τους πολίτες της Ευρώπης. Πολύ συχνά πολίτες στη δική μου περιφέρεια ε, μου λένε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα, γιατί υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίοι παίρνουν τους ευρωπαϊκούς χώρους, πόρους, αλλά από την άλλη δεν τηρούν τους κανόνες παιχνιδιού και περιφρονούν τις δημοκρατικές αξίες. Μία λειτουργία του κράτους δικαίου είναι ουσιαστική, ε, καθοριστική για μια καλή ε, χρησιμοποίηση των πόρων. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος της ε, απάτης. Γι' αυτό είναι σωστό να εκπονήσουμε αυτό το εργαλείο. Αλλά όχι δικαιούχοι, οι φοιτητές, οι γεωργοί θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες, αλλά οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θέλουμε ε, κυρώσεις για χώρες οι οποίες ε, χρησιμοποιούν ε, αθέμητα φορολογικά συστήματα. Εάν θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή οικογένεια, τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον προστατεύουμε τις δημοκρατικές μας αξίες και να χωρίς αντιπαραθέσεις μεταξύ μα αλλά συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κοινό προπολογισμό είναι η ρεχοκαλιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δράσει στην αρχή τη αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρέ οικονομικά χώρε είναι διατεθειμένε να αναλάβουν ε, ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη. Άρα είναι προφανές ότι η εφομείωση των πόρων θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Ε, Αλλιώς η αρχή της αλληλεγγύης ε, δεν οδηγεί πουθενά. Το κράτος δικαίου είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κρότες, ε, τα κράτη-μέλη ε, είναι υποχρεωμένα να τηρούν αυτές τις αρχές. Εάν μια χώρα συστηματικά παραβιάζει αυτές τις αρχές, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε παρκώς. Γι' αυτό στηρίζουμε αυτό το νέο μηχανισμό και ευχαριστούμε την Επιτροπή για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας. Ιδιαίτερο σημαντικό σημαντικό είναι για μας μια μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού ε, γιατί είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες. Προχωρούμε στη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι ορισμένοι ομιλητέ φοβούνται την κατάχρηση αυτού του προτινόμενου κανονισμού. Ναι, όπως και κάποιοι πρωθυπουργοί καταχρώνται τις θέσεις τους και ο κίνδυνος αυτός υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω όμως πως οι αρχές της Ένωσης θα πρέπει να προστατευτούν τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν υπάρχει κατάχρηση θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία στη διάθεσή μας ώστε να ε, διορθώσουμε την κατάσταση. Αρκετές φορές ε, έχουμε μιλήσει για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 και, και έχουμε ψηφίσει συγγνώμη, για την ενεργοποίηση του 7 και εγώ ποτέ δεν το υπερψήφισα διότι αυτό στιγματίζει μια κυβέρνηση. Βλέπουμε επίσης πως αυτό το εργαλείο δεν αρκεί για να προστατέψει τον προπολογισμό της Ένωσης και το κράτος δικαίου. Χρειαζόμαστε καλύτερο αμυντικό μηχανισμό και σας ευχαριστώ. για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, διάβασα προσεκτικά αυτή την έκθεση η οποία μου θυμίζει το βιβλίο του George Orwell. Οι Ευρωπαίοι κάθε μέρα γίνονται μια αληθινή φάρμα, όπως το βιβλίο του Orwell. Ορισμένες, κράτες, ε, ορισμένες χώρες είναι πιο ίσες από άλλες. Στην έκθεση γίνεται κατά επανάληψη αφορά, αναφορά σε το μηχανισμό διόρθωσης. Ωστόσο δεν υπάρχουν παρά μόνο δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες εφαρμόζεται αυτός ο μηχανισμός. Κύριε Πίτροπε, ε, αν θέλ, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση, θα πρέπει πριν από αυτό όλες οι χώρες ε, μέλη να υπόκεινται σε αυτόν τον μηχανισμό. Εφαρμόστε αυτή την πρακτική στις δικές σας χώρες, αλλιώς δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των χωρών. Η αρχή της προστασίας των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί μεν να είναι δικαιολογημένη, αλλά η διαδικασία με ανησυχεί. Διαβάζοντας αυτή την έκθεση είχα την αίσθηση ότι θέλει να μας ε, φοβήσει. Ε, να μας φοβήσει λέγοντας ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να μείνουμε μάδια στις τσέπες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι η Επιτροπή αυτή η οποία καλείται να αναγνωρίσει, τις, να ανοιχνεύσει και να εντοπίσει τις γενικευμένες ελλείψεις στη βάση όλων των διαθέσιμων πηγών ε, που έχει στη διάθεσή της. Ποιες είναι αυτές οι πηγές, είναι τα ΜΜΕ, είναι η ΜΚΟ, είναι οι καλοπροαίρετοι συνάδελφοι από άλλες χώρες. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ψηφίζουμε τέτοιου είδους πράγματα. Ευχαριστώ. Δείτε το χρόνο του ΚΑΤΣΤΙΑ για να μιλήσουν όλοι. Ε, ο κύριος Μαριάς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το άρθρο 7 προσδιορίζει την προστασία του κράτους δικαίου και βεβαίως των αξιών της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά η λειτουργία του άρθρου 7 γίνεται εντός του πλαισίου λειτουργίας της ίδιας συνθήκης δηλαδή οφείλει η εφαρμογή του άρθρου 7 να σέβεται τις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής ένωσης. επομένως το άρθρο αυτό θα λειτουργεί στο πεδίο όπου υπάρχει αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής ένωσης και όχι εκτός βεβαίω όλοι θέλουμε να χτυπηθούν οι απάτες και αυτό είναι δεδομένο. δεν πρέπει όμως να αξιοποιείται το άρθρο 7 και ο μηχανισμός ο οποίος προτείνεται ως ένα πολιτικό εργαλείο επέμβασης στα εσωτερικά των κρατών και να εκφράζεται έτσι επί της ουσίας μια νέο-απικιακή πολιτική. υπάρχει και διγλωσία όταν η τρόικα και οι μνημονιακές κυβερνήσεις στην ελλάδα παραβίαζαν το κράτος δικαίου και αυτό το καταγγείλαμε επανειλημμένα εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν είδαμε να λαμβάνονται μέτρα. αντίθετα μας είπαν ότι η εφαρμογή των μνημονίων παρότι παραβίαζε τα θεμελιώδη δικαιώματα ήταν νόμιμη. πρέπει λοιπόν να προσέξουμε για το πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός. ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ε, αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι πολύ σημαντική και δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι ε, αυτό είναι το αντικείμενο της πρότασης για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης η προστασία όλων μας δεν μπορεί να συνδεθεί με τους πόρους των διαφόρων κρατών μελών, διότι αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση παραβάσεων και της κακής λειτουργίας του δικαστικού συστήματος ε, θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, σε, κάποια κράτη-μέλη ενώ θα επιβάλλονται λιγότερες κυρώσεις σε κράτη-μέλη που λαμβάνουν ε, λιγότερους πόρους. Ενώ έχουμε βελτιώσει σημαντικά την πρόταση αυτή, θα πρέπει να την βελτιώσουμε περαιτέρω για να διασφαλίσουμε την ενιαία εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη άσχετα από τους πόρους που λαμβάνουν domnule președinte stimați colegi bugetul uniunii europene este extrem de important pentru fiecare cetățean al statelor membre. Είναι πολύ σημαντικός ο προϋπολογισμός για τους Ευρωπαίους. Υποστηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης. Και στη δική μου χώρα έχει βοηθήσει ο προϋπολογισμός, όπως και τα ταμεία. Απασχόληση, εξυγχρονισμός, υγεία. Άρα θέλουμε όλοι να αξιοποιούνται οι πόροι για το όφελος όλων. Θέλουμε να υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος επί του προϋπολογισμού, αλλά τα πολιτικά κριτήρια για τις κυρώσεις είναι ένα μέτρο το οποίο περικλεί κινδύνους να αποφύγουμε την περίπτωση του να χειραγωγείται ένα κράτος ή τέλο πάντων να γίνει παιχνιδάκι για μικροπολιτική. Θέλουμε να υπάρχει ρύθμιση δίκαιη, ισοτιμία, να μην έχουμε αμφιβολίες. Ε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Έτιγκερ. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία ελέγχθησαν, θα τα αξιολογήσουμε και θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία έτσι ώστε η δυνατόν ε, να υπάρξει μια καλύτερη επεξεργασία της πρότασής μας, η οποία είναι και η βάση ε, της νομοθεσίας. Από τις ε, απόψεις που εκφράστηκαν βλέπω συνεπέραν ότι οι περισσότεροι συμφωνούν με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιθυμούν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι αν θέλουμε το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει όλες οι διαδικασίες να είναι νομότυπες και στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία αυθαιρεσία ούτε καν κομματική προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν στην πρόταση Επιτροπής καθορίσαμε το πώς πρέπει να εργαζόμεθα, πώς πρέπει να διαφυλάσσουμε την αντικειμενικότητα, να ε, αποκλείουμε παρεμβάσεις. Ε, ε, καταλάβαμε πώς πρέπει να αιτιολογούμε τις προτάσεις μας. Εξάλλου, το θυγόμενο κράτος μέρος ε, ή μέλος, με θα πρέπει να εισακούεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι η μόνη η οποία φέρει την ευθύνη. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ε, το Συμβούλιο μπορεί να αναπέμψει προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν τελικά ε, λουφθεί μία απόφαση, η απόφαση αυτή ε, πρέπει να εφαρμόζεται και μπορεί να αμφισβητηθεί σε δικαστήριο αν κάποιο κράτος μέλος αισθάνεται ότι φύγεται. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει ε, πράγματι να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις των δικαστηρίων τα οποία θα είναι και καθοριστικά για το μέλλον και για τις προσακολουθούμενες διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωρούμε στους ε, εισηγητές. Η κυρία Γκάρια Θάμπαλ Ρουμπιάλ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Δεν θα αργήσω. Ήταν μεγάλη ημέρα και ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας στην Σύνοδο. Πάντως, σε σχέση με αυτά που είπε ο Επίτροπος, άκουσα όσα συζητήθηκαν άκουσα τις θεμητές αμφιβολίες και επιφυλάξεις και ο κύριος Σαρβαμά και εγώ θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας θα απασχίσουμε για μια συμφωνία με την Ρουμανική Προεδρία οπότε να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Σαρβαμά για τη συνεργασία ξεκινήσαμε από κάπως θέσεις που ήταν σε απόκληση αλλά τελικά μια καλή έκθεση έτσι φτιάχνεται και επίσης βοήθησαν και οι διαπραγματευτές όλων των πολιτικών ομάδων η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και η Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο και τους συνεργάτες του. Όλοι συνέβαλαν απλώς. Ελπίζω ότι αυτά που διαπραγματευτήκαμε τους τελευταίους ε, μήνες θα επικυρωθούν με την αυριανή ψήφο. Θα πάμε για διαπραγματεύσεις και θα φτιάξουμε ακόμα καλύτερο το κείμενο. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο εξηγητής ο κύριος Σάρβαμα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλες τις παρεμβάσεις. Θα ήθελα να ακολουθήσω μία κάπως συνήθιστη σειρά, δηλαδή να σας ευχαριστήσω καταρχήν και μετά να πω τις τελικές παρατηρήσεις. Όσους δεν ευχαρίστησα στην αρχή, τους ευχαριστώ τώρα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους όσους συνεργάστηκαν, τους κοιόδης εισηγητές, τις γραμματείες, ε, εξαιρετικοί συνεργάτες σε όλες τις επιτροπές. Αλλά κάτι που θέλω να πω πριν πω και το κλείσιμο της παρέμβασής μου, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτούς που ακολούθησαν επικοδομητική στάση. Ίσως που δεν ενέκριναν απολύτως την έκθεση ή την πρόταση, αλλά ήταν πολύ επικοδομητικοί. Με κάποιες επιφυλάξεις, με κάποιες ιδέες για τις τριμερείς συζητήσεις. Και τέλος, κλείνοντας, Θέλω να πω ότι ε, νιώθω πολύ απογοητευμένος, διότι έτσι δουλεύει η πολιτική. Ακούσαμε απόψε πολλούς ομιλητές που δεν ήταν έντιμοι. Μιλούσαν βασικά στο εθνικό τους ακροατήριο. Και αυτό πρέπει να το πω. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια παρατηρούμε την τραγική φάρσα των πολύ σημαντικών συνεπειών που έχει αυτή η πολιτική για ένα μεγάλο κράτος και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Και δυστυχώς μερικές φορές αυτό είναι η πολιτική. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δουλέψουμε ειλικρινά για μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ έληξε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ με θέμα τη θέσπιση του προγράμματος Φισκάλης για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Εξ του εισηγητή, το λόγο έχει για τέσσερα λεπτά η συνάδελφος Σκοτ Κάτου. Thank you very much, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Έτιγκερ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και οικονομικού εγκλήματος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από κάθε χώρα μόνη τη λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα τη απάτης. Η αυξημένη συνεργασία λοιπόν και μια πραγματικά ευρωπαϊκή ε, απάντηση στην φοροαποφυγή είναι απαραίτητη. Δυστυχώ στο Συμβούλιο οι κυβερνήσει μπλοκάρουν βασικά νομοθετικά κείμενα που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά και που θα μπορούσαν να κάνουν τις μεγάλες εταιρείες και τα πλούσια άτομα να πληρώσουν το μερίδιό τους και όσον αφορά την κοινή βάση φορολογίας και όσον αφορά άλλες φορολογικές διατάξεις. Χθε ε, προτάθηκε να περάσουμε στην ε, ε, πλειοψηφία και να δοθεί στο Κοινοβούλιο μεγαλύτερη δραστηριότητα. Όμως η Επιτροπή επέλεξε λάθος εργαλείο για να επιτύχει το στόχο. Γιατί υπάρχει μια μη αποτελεσματική ρήτρα πασαρέλα αντί να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 116. Ωστόσο, δεν είναι υπεύθυνη η Επιτροπή, αλλά τα κράτη-μέλη για αυτή